και κύριοι, περνάμε στην ψηφοφορία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος μέχρι την ε, εκδήλωση που έχουμε σε 15 λεπτά από τώρα την παρηγενική συνεδρίαση και το υπόλοιπο θα έρθει μετά. Λοιπόν, ε, πολιτική συνοχή υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε στην έκθεση για την με Ομάριε. Βελτιστοποίηση ανάπτυξη του δυναμικού των εξόχων από και των περιοχών. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην έκθεση. Ορίστε. Έκθεση Τόιρερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έκθεση Ντεμπάκερ. Τον λόγο έχει ο εισηγητής. Κύριε Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ. Ε, από πλευρά τη Άλντε θέλω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για σήμερα ε, και για αυτήν την ε, σύνοδο σύμφωνα με την διάταξη 177 του καταστατικού. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματος αναβολής? Ποιος θα μιλήσει υπέρ? Θέλει κάποιος να μιλήσει κατά? Κανείς. Περνάμε στην ψηφοφορία. Υπέρ της αναβολής. Κατά. Αποχές. Ωραία, το έτοιμο γίνεται δεκτό. Οπότε περνάμε στην έκθεση Σαλαφράγκα, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην έκθεση Βέμπερ, Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας ε, με Κώστα Ρίκα και λοιπές χώρες. Υπέρ, κατά αποχές δεκτή έκθεση Μπερές ονομαστική ψηφοφορία άρχιτη ψηφοφορία πέρασε δεκτή περνάμε στην έκθεση για το κοινό σύστημα ΦΠΑ, straight check. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην έκθεση Hübner. Ονομαστική ψηφοφορία υπέρ. Ε, με συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Δεύτερη έκθεση της κυρίας Χίμπνερ για την Μαγιότ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Έκθεση της κυρίας Άννα Γκόμες υπέρ της έκθεσης με ανατάσσεω χειρός κατά αποχές εγκρίνεται η έκθεση περνάμε στην επόμενη έκθεση της κυρίας Γκόμες υπέρ κατά αποχές δεκτή Άλλη μια έκθεση της κυρίας Γκόμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Επόμενη έκθεση της κυρίας Ρενάτα Ζόμερ. Για τη συμφωνία με την Τουρκία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε. Ορίστε κύριε συνάδελφε. Κύριε Κάλαχαν. Η επόμενη ψηφοφορία για την παράταση του άρθρου 147. Θα ήθελα να ζητήσω από τους βουλευτές να καταψηφίσουν γιατί πρόκειται για άλλη μια επίθεση κατά της Ιρλανδικής γλώσσας. Mm. Νομίζω πως είναι ανετιολόγητος ο φόβος σας. Περνάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Η κυρία Ρούσα Τόμασακ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε διδάξει 146 παραγωγή 1 και 2. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, είμαι θα κατά της πρότασης ούτως ώστε να επεκταθεί η ισχύση του 147 όσον αφορά ε, στην ε, καθυστέρηση της ε, χρήσης ή στο, των κροατικών στις εργασίες μας. Είναι επίσημη γλώσσα και θα πρέπει να μην θεωρείται γλώσσα δεύτερης κατηγορίας. Δεν δέχομαι την παρούσα γιατί ένα χρόνο αφού η Κροατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι να συγκροθεί σε σώμα το επόμενο κοινοβούλιο, μέχρι τότε ε, υπάρχει αρκετός χρόνος τόσο ώστε να υπάρξει πλήρης κάλυψη όσον αφορά την κρατική γλώσσα. Όπως είπα τα έχουμε εξετάσει όλα αυτά στο Προεδρείο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην έκθεση Καζίνη. Τροπολογία 3 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 1 καταπίπτει. Ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2 καταπίπτει. Περνάμε στο στο σύνολο της έκθεσης με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εκτή. Έκθεση ε, Ελχαντραουή για τον ε, Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Φόρο έχουμε 68 τροπολογίες με αναψυχή ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 5 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 9. Διανατάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 32 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε. Τροπολογία 37 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε. απορρίπτεται τροπολογία 47 πάλι σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 47 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 80 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 51-91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 93 έως 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 96. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 57 καταπίπτει. Ήταν, ήταν σαφές. Τροπολογία 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεχτεί. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η επόμενη καταπίπτει όχι 123 CP υπέρ κατά εποχές δεκτή 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή 101 και 125 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεκτή να την επαληθεύσουμε αρκετή ψηφοφορία πέρασε Απορρίπτεται. Οπότε σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 της Επιτροπής υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ τρίτο μας κατά αποχές δεκτή 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή 106 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 82 της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές δεκτή 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ κατά αποχές δεκτή 109 υπέρ κατά αποχές δεκτή 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές δεκτή να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές δεκτή 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στην ψηφοφορία επί της πρώτης κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή. Περνάμε στο νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συγχαίρω τους εισηγητές. Η συνεδρίαση διακόπτεται μέχρι τις 12.30 και για την ομιλία του Προέδρου της Τσεχικής Δημοκρατίας.